So, ladies and gentlemen. Ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να καθίσετε. Please. It's necessary to continue. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε δουλειά ακόμα. So if you allow me, I would like... Λοιπόν, άμα επιτρέψετε θα μιλήσω σλοβακικά σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ε, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Επιτρέψτε μου να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της Προέδρου κυρία Βίξτρομ ε, που δυστυχώς κολλείται και δεν μπόρεσε να φτάσει στις Βρυξέλλες λόγω καιρού. Είχε πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Ελπίζω να φτάσει αργότερα. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Έχετε να κάνετε σχόλια, παρατηρήσεις στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν έτσι η μερική διαταξή. Δεύτερο σημείο. Έγκριση του σχεδίου μερικής διάταξης. Μάλλον όχι, αυτό το εγκρίναμε. Είναι το 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 22-23 Νοεμβρίου και 28 Νοεμβρίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχετε παρατηρήσεις να κάνετε σχετικά με τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών. Όχι. Ωραία. Εγκρίνονται λοιπόν και τα πρακτικά. Πριν συνεχίσουμε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρία των συντονιστών προηγουμένως διεκόπη δεν ολοκληρώθηκε. Θα υπάρξει και συνέχεια αύριο διότι είχαμε κάποια προβλήματα να συζητήσουμε που χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Οπότε θα ε, αναβληθούν αυτά για αύριο και επίση θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά από τη σημερινή συνεδρία έχουμε μια μικρή δεξίωση πρωτοχρονιάτικη κάτω στο ισόγειο, στα σαλόνια των βουλευτών, όπου είστε προσκεκλημένοι θερμά όλοι. Και τώρα ακολουθεί ε, η ε, κανονική εργασία της Επιτροπής μας. Περνάμε στις αναφορές προς συζήτηση. Έχουμε το σημείο 6, αναφορά αριθμός 1498, κάθετος 216. Έχει υποβληθεί από τον κύριο Όρος, Σλοβάκο πολίτη, ε, έχει να κάνει με τη βιότητα ε, του πόσιμου ύδατος ε, στην συνοικία Βράκουνια ε, της Μπρατισλάβα. Επειδή είναι παρόν αναφέρον, θα ήθελα να του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές για την πολύ ευγενική τους πρόσκληση που με κάλεσαν να εξηγήσω εδώ αυτήν την ε, αναφορά. Βρίσκομαι εδώ εκ μέρους των πολιτών που ζουν σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο νησί του Δούναβη στην Νότια Σλοβακία. μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την Αυστρία, μόλις 10-20 χιλιόμετρα, ε, στα σύνορα πάνω με την Ουγγαρία. Η Βρακούνια είναι κομμάτι της ε, Μπρατισλάβα. Το νησί αυτό ε, χτίστηκε, κατασκευάστηκε μάλλον μέσα σε πολλές χιλιατηρίδες από τον ίδιο το Δούναβη. και κάτω από αυτό το νησί. Έχουμε τεράστια αποθέματα γλυκού νερού. Δυστυχώς, για εδώ και δεκαετίες, ε, το εργοστάσιο χημικών προϊόντων Δημητρόφ αποθηκεύει επικίνδυνα απόβλητα στο νησί αυτό. Αφού χτίστηκε το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Χαπκατσίκοβο, ε, έχει δημιουργηθεί μια ανεύθυνα κατασκευασμένη χωματερή. Μια αυθαίρετη χωματερή και έχουμε 90.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων που μετά από κάποια ζημιά διαραίουν στο έδαφος. κινούνται προς τα δυτικά κατά 600 μέτρα ετησίως και τώρα ρηπαίνουν ε, τοπικά πηγάδια Η χρήση ε, των τοπικών πηγαδιών έχει απογρευτεί μετά από το 2002 διότι τα ύδατα είναι επικίνδυνα ειδικότερα για τα παιδιά. Εδώ βλέπετε ένα χαρτί υψηλής ανάλυσης ε, όπου βλέπετε την περιεκτικότητα της ρήπανση 5, 10 και 15 μικρογραμμαρίων. Εδώ βλέπετε την έκταση ουσιαστικά της ρήπανση της ζημιάς. Εδώ βλέπετε την περιοχή όπου έχουν θαυτεί τα βαρέλια. Πριν από τα Χριστούγεννα τεκμηριώθηκε και άλλη μία πηγή ρήπανσης παρότι η ακριβής πηγή δεν είναι γνωστή. Χρειάστηκε να φέρουμε πόσιμο νερό, διότι το τοπικό νερό έχει ρηπανθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Έχει κατασταθεί εξοπλισμό ε, φιλτραρίσματος, ωστόσο το έδαφος παραμένει μολυσμένο. Το Υπουργείο έχει κάνει διάφορες υποσχέσεις, οι μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν ότι η μολυσμένη περιοχή θα ε, περιοριστεί. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία ανθρώπων σε μια δράση διαμαρτυρίας κατά της αδράνειας των αρχών. Το σχέδιο είναι ουσιαστικά να κατασκευαστεί ένας ε, τείχος βάθους 20 μέτρων ε, σε περιοχή 2 χιλιόμετρων με κόστος 13 ε, εκατομμύρια ευρώ. Θα κατασκευαστεί ο τείχος αυτός από σκυρόδεμα. και θα αντιστοιχεί στο 1 τέταρτο του κόστους απόσυρσης των βαραλιών και εξουδετέρως της των τοξικών αποβλήτων. Αυτή η απόφαση λοιπόν που προτίμησαν οι τοπικές αρχές δεν είναι ιδανική. Αυτό που προτείνω εγώ και αυτή δεν είναι η τελική μου πρόταση αλλά αυτό που προτείνω είναι να διατηρήσετε την ε, αναφορά αυτή ανοιχτή είναι πιθανό να επηρεάσει και μια από τις πρωτεύουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς και τρεις συνολικά χώρες η λύση που προτείνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι παραπροσωρινή. Υπολογίζω λοιπόν στην βοήθειά σας και στην προσοχή που ελπίζω να δώσετε στο μέλλον. Ελπίζω ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να δώσουμε τέλος σε αυτή τη μόλυνση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από ευκαιρία να ζητήσω συγγνώμη ε, που καθυστέρησα τόσο πολύ. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί και ήταν αδύνατο να αναχωρήσει οτιδήποτε δεν μας έδιναν άδεια να πετάξουμε και περιμέναμε και περιμέναμε και κάποια στιγμή προσγειώθηκα στο Μόναχο και που είχε έλα και δεν μπορούσε ο πιλότος να προσγειωθεί. Κάναμε βόλτες πάνω από το Μόναχο πάρα πολύ ώρα και έχασα την ανταπόκριση. Αλλά σας ήρθα πάντως ε, υγιής και διάθετη όλα αυτά. Ελπίζω να ε, μοιραστούμε αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά. Με ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το σωτήρα μου, τον κύριο Σάκη, ο οποίος πάντα είναι ο καλύτερος συνάδελφος. Έρχεται, αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, προεδρεύει και σέβεται και μάλλον ε, σώνει τη δουλειά της Επιτροπής. Πραγματικά έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και ελπίζω και κάποια στιγμή να ε, ανταμευθείτε στον παράδεισο για αυτά που κάνετε εδώ στη γη. Λοιπόν, προχωρούμε. Και το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η κυρία Βοχέμοβα. hello, good afternoon. Καλησπέρα σας. Εδώ εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση για να γνωρίζετε κι εσείς για το τι συμβαίνει με αυτή την αναφορά. Να προσθέσω στα όσα σας στείλαμε τον Ιούνιο, να σας πω πως τον Οκτώβριο ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές στην Πρατισλάβα και συζητήσαμε και το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που είναι η αποκατάσταση ε, της περιοχής Βρακούνια, και το Υπουργείο στη Σλοβακία μας είπαν πως αποδίδουν τη μέγιστη προτεραιότητα έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η χωματεροί και μας προσέφεραν μάλιστα και ένα χρονοδιάγραμμα και μας είπαν πως θα ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα σε έξι μήνες. Εν τω μεταξύ όμως σημειώθηκε κάποια ακόμα καθυστέρηση οπότε το Δεκέμβριο μας έστειλαν και ένα επόμενο χρονοδιάγραμμα και μας είπαν πως κανονικά θα πρέπει η χωροθέτηση και η άδεια για τη χωροθέτηση να έχει δοθεί το Μάρτιο έτσι ώστε το Δεκέμβριο του 2018 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Βέβαια με την επιφύλαξη και κάποιων άλλων καθυστερήσεων. Αυτό που είναι θετικό είναι πως το θέμα των κρατικών ενισχύσεων έκλεισε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της Σλοβακίας και μπορεί αυτή τη στιγμή να λάβει και οικονομική στήριξη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ποιότητα περιβάλλοντος κάποια κονδύλια. Λοιπόν, από το πρόγραμμα αυτό θα διατεθούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εξετάζει το πρόγραμμα για τη διαχείριση των ε, ε, ποταμών όλων των κρατών μελών και μέχρι τα τέλη του 2018 θα σας παρουσιάσουμε τις σχετικές πληροφορίες και αντιμετωπίζουμε κυρίως κάποια συστημικά θέματα που έχουν προκύψει. Τέλος, να σας πω πως δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθεί την αποκατάσταση, ούτε να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή. Είναι θέμα που πρέπει να αποφασιστεί σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Οι συνάδελφοι τώρα έχουν το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Στέφανεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου κι εγώ. ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συντάκτες της αναφοράς. Πραγματικά πρόκειται για το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής εκεί, ρηπαίνεται το περιβάλλον και η κατάσταση πλέον είναι αφόρητη. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, ε, χρονίζει και μάλιστα μέσα σε γενική αδιαφορία. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα οι πολίτες υψώνουν τη φωνή τους και καταθέτουν τη συγκεκριμένη αναφορά. Αυτή η χωματερή εκεί έχει τοξικά απόβλητα και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και κίνδυνος για το περιβάλλον, όχι μόνο για τη Βρακούνια ή άλλες συνοικίες της Βρατισλάβας, αλλά και για άλλους δήμους και γειτονικού ε, σε αυτό το μεγάλο νησί στο Δούναβι. Δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί μόνιμα, όχι με εμβολωματικές λύσεις για το σημερινό πρόβλημα. Μια συνολική λύση χρειάζεται. Άρα, ε, πρέπει να αναζητήσουμε μακροχρόνιες λύσεις. Γι' αυτό θα χαιρόμουν αν η κατάσταση αυτή και η αναφορά αυτή παρέμενε ε, ανοιχτή και είναι κάτι που να το εξετάζει μακροχρόνια και μακροπρόθεσμα και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ πάλι. Θα μιλήσω και εγώ σλοβακικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και επίσης να ενημερώσω την Επιτροπή ότι αύριο θα έχουμε ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους σοσιαλιστές και άλλους βουλευτές μη εγγεγραμμένους που θα ε, ζητούμε από κοινού από τη Σλοβακική κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί επιγόντως. Είναι πάρα πολύ καυτό το ζήτημα, πάρα πολύ επίγον και χρειάζεται ταχύτατη ε, δράση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι πάρα πολύ κοντά στα υπόγεια ε, ύδατα και στον υδροφόρο ορίζοντα αυτή η χωματερή υπόγεια και κινδυνεύει ε, να ρηπάνει όλο το νερό της Μπρατισλάβας πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Μήπως ε, θα ήταν καλό να στείλουμε και επιστολή στη Σλοβακική κυβέρνηση και να την καλούμε να βρει μια λύση το συντομότερο. Ε, είναι ο ορίζοντα ορίζοντας τη της τη Πρωτισλάβα. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε για το τι θα πρέπει να γίνει με την αναφορά αυτή παραμένει ανοιχτή και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη και πιο πλήρη αξιολόγηση κατάσταση αργότερα. Εν τω μεταξύ θα στείλουμε μια επιτροπή στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Σλοβακία και θα τους ρωτήσουμε τι ακριβώς κάνουν οι αρχές στη χώρα για να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα πλαίσια αυτής της αναφοράς και επίσης μια λεπτομερή εξήγηση για το τι σχεδιάζουν και τι συνέχεια θα δώσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά τα οποία οι αναφέροντες μας υποβάλλουν. Θα ήθελα να επαναλάβω πως εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα της χρήσιμης αναφοράς, όχι μόνο για τη Σλοβακία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις χώρες οι οποίες επηρεάζονται από το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν εμπίπτει απολύτως στο πεδίο αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών οργάνων και νομίζω ότι είναι και μια επίγουσα αναφορά λόγω του θέματος. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι σε εσάς. Είχα ξεχάσει σχεδόν πως πρέπει ο αναφερόμενος να ξαναλάβει το λόγο και να συμφωνήσει ενδεχομένως μαζί μου πως είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Στέφανε, ο οποίος με βοήθησε και με στήριξε και επίσης και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πάσκη, για τη στήριξη που προσφέρει. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πως παρόλο που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τη λύση και πως παρόλο που έχει κάνει κάποια βήματα η Σλοβακική κυβέρνηση, πρέπει να σας πω ότι έχουν περάσει 14-15 χρόνια με διαμαρτυρίες, καταγγελίες του τοπικού πληθυσμού και επιτέλους κάτι γίνεται. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε εκατοντάδες κυβικά μέτρα τσιμέντου που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για να χτιστεί ένα τείχο στη μέση του νησιού μας. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη δυνατόν λύση. Και να σας πω επίσης πως τα έξοδα και οι δαπάνες για τη λύση αυτή είναι συγκρίσιμα με μια τελική λύση που θα μπορούσε να δοθεί και η οποία βέβαια θα κόζει τέσσερις φορές παραπάνω από αυτό τον ε, τείχο προσκυρόδεμα και θα αποτελούσε και μια τελική λύση. Οπότε θα ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βρει τους πόρους για να στηρίξει τη σλοβακική κυβέρνηση και να αποκατασταθεί η ευρύτερη περιοχή Χαίρομαι λοιπόν που συμφωνήσατε μαζί μου και θα ακολουθήσουμε αυτά τα οποία πρότεινα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι αντίθετο. Όχι. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που το πολύ σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό θέμα το αναφέρατε στην καρδιά της Ευρώπης που είναι οι Βρυξέλλες. Και σας εύχομαι και καλή επιστροφή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η αναφορά 1497 του 2016. Είναι ο Παναγιώτης Λελιάτσος που μιλάει για τις καταχρηστικές διατραπεζικές προμήθειες, ηλεκτρονικές συναλλαγές που επιβάλλονται. Να ένα θέμα. Ο αναφερόμενος βρίσκεται εδώ. Είστε εδώ. Όχι. Άρα λοιπόν θα δώσω απευθείας το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα. Ε, έρχομαι από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής. Η αναφορά ουσιαστικά αναφέρει δύο στοιχεία. Ένα επί της ουσίας και ένα διαδικαστικό σε σχέση με την ε, διακυβέρνηση. Ας σας μιλήσω πρώτα για το επιχείρημα επί της ουσίας. Ε, ισχυρίζεται ο αναφέρον ότι ως αποτέλεσμα της ελληνικής νομοθεσίας Όσον αφορά τα capital controls, ε, η, χρέωση, η χρήση μάλλον των ε, τραπεζικών και επιστοτικών καρτών έχει αυξηθεί και ενδεχομένως το αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες χρεώνουν ε, στους εμπόρους τέλη που ανέρχονται έως και στο 3% της συναλλαγής. Ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι αυτό αποτελεί παραβίαση αυτού που ουσιαστικά ε, έχουμε ρυθμίσει στον κανονισμό για τα σχετικά τέλη. Εμείς ε, στις παρατηρήσεις μας έχουμε αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που υπησέρχονται τα συστήματα καρτών πληρωμών. Ε, είναι ένα περίπλοκο δίκτυο σχέσεων μεταξύ πολλών παραγόντων και εφαρμόζονται διάφορα τέλη ο σχετικός κανονισμός αριθμίζει μόνο ένα στοιχείο όλων αυτών, τα τέλη τα οποία χρεώνουν ε, οι τράπεζες οι οποίες εκδίδουν ε, ε, κάρτες και το ανώτερο όριο που εφαρμόζεται εκεί. Τώρα για τις πληρωμές με κάρτες επιβάλλονται περαιτέρω τέλη από κάποιες ε, τράπεζες ε, στους εμπόρους και ε, τελικά στον τελικό καταναλωτή. Εδώ είναι και το πρόβλημα εδώ, διότι κάποια από αυτά τα τέλη μπορεί να υπερβαίνουν αυτές τις οροφές, αυτά τα ανώτερα όρια που έχουμε ρυθμίσει εμείς, αλλά αυτά τα επιπλέον τέλη δεν αποτελούν το αντικείμενο ρύθμισης. Τα κρατη λοιπόν και οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις τα ρυθμίζουν αυτά τα τέλη βάσει της αγοράς. Αυτό σχετίζεται με το τι συνήθως χρεώνονται στους εμπόρους που ονομάζεται τέλος χρέωσης εμπόρου που αποτελείται από, αυτούς τους ρυθμιζό, από αυτά τα ρυθμιζόμενα τέλη συναλλαγή ε, και από άλλα τέλη που μπορεί να επιβληθούν για διάφορου λόγου. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα διαφόρων άλλων τελών που επιβάλλονται ε, διάφορων ειδών ε, τελών διεκπαιρέωση. Ε, υπάρχουν διάφορα, πολλά διαφορετικά τέλη που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως. Ε, το θέμα είναι τώρα ότι οι τράπεζες, οι εκδοτικές τράπεζες μπορούν να επιβάλλουν τέλη στους εμπόρους που να υπερβαίνουν ε, τα αριθμιζόμενα τέλη. Συνήθως δεν φτάνουν σε τόσο μεγάλα ποσοστά 3% περισσότερο κοντά στα τέλη που έχουμε ρυθμίσει εμείς τα, τα τέλη των συναλλαγών αλλά αυτό που μπορούμε εμείς να πούμε εδώ ε, γιατί μπορούμε να σα εξηγήσουμε μόνο το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί δεν ξέρουμε σε τι ακριβώ αναφέρεται ο αναφέρον. Μπορεί να είναι το ζήτημα των εμπορικών καρτών που δεν καλύπτονται από το ε, κανονισμό, όπου τα τέλη είναι πολύ ψηλά, πολύ κατά πολύ ψηλότερα. Πολλά στοιχεία λοιπόν τελών ε, χρεώνονται στους εμπόρου ενδεχομένω και που είναι μεγαλύτερα από τα ρυθμιζόμενα τέλη. τραπεζικές, ε, αυτά τα τραπεζικά τέλη λοιπόν που μπορεί να είναι και παραπάνω από 3% κάτι που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό αυτό είχα να πω όσον αφορά την ουσία, όσον αφορά τα τέλη. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο της αναφοράς ε, για το οποίο διαβουλευτήκαμε τις ελληνικές αρχές. Αυτό σχετίζεται με τον ορισμό αρμοδίων αρχών που επιτηρούν την εφαρμογή του κανονισμού διατραπεζικών τελών. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ελληνικές αρχές μας απάντησαν λέγοντας μας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, ο δεσμευτικός στόχος του κανονισμού, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική υποπτική αρχή. Δεν χρειάζεται να είναι μια νέα αρχή, μπορεί να, να είναι και μια υπάρχουσα αρχή ε, στην οποία θα ανατεθεί το έργο αυτό βασικό των πληροφοριών που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απόφαση ποιος θα αναλάβει δηλαδή στην Ελλάδα αυτό το έργο. Μας ενημερωσαν ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει έρθει σε επαφή με πολλές εθνικές ε, αρχές όσον αφορά αυτή τη δέσμευση, το Υπουργείο Οικονομίας, την ε, Τράπεζα της Ελλάδος, τον Έλληνα Δημοσιολαβητή και την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού. Το Συνήγορο του Πολίτη Μόλις θα λάβουμε λοιπόν τις σχετικές πληροφορίες θα σας ε, ενημερώσουμε για το πώς πρόκειται να, ε, από ποιον πρόκειται να αναλυθεί αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η υποχρέωση. Ευχαριστώ. Okay. I... Ωραία, ευχαριστούμε. Όπως κατάλαβα η ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Κάτι πολύ καλό. Διότι δεν έχει νόημα απλά να περιμένουμε και να αναβάλουμε μια ε, απόφαση απόφαση που θα μας πει ποιος είναι αρμόδιος. Δεν ξέρω τι περιμένουν οι ελληνικές αρχές για να λάβουν μια απόφαση. Περιμένουν εδώ και μήνες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που μας ξεκαθάρισε κάπως την κατάσταση και που συνεχίζει να την παρακολουθεί, ε, επιδιώκει να βρεθεί μια λύση, συνεργάζεται μαζί μας για να βρούμε μια λύση. Ευχαριστούμε λοιπόν για την πολύ ε, πλήρη περιγραφή αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Ε, λυπάμαι που αποφάσισε να μην έρθει ο αναφέρον, διότι είναι πολύ καλή αναφορά αυτή. Θα ήταν πολύ καλό να ήταν εδώ ο αναφέρον. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αναφορά. Εμείς συζητήσαμε ο CCR να επισπευθεί η συζήτησή της και να έρθει στη σημερινή ημερήσια διάταξη διότι το θέμα της καταχρηστικής λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα είναι στην ημερήσια διάταξη. Όσον αφορά το διαδικαστικό μέρος το οποίο αναφέρθηκε η Κομισιόν και πολύ σωστά αναφερθήκατε κι εσείς, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση όταν έχει απαιτήσει από την Τρόικα νομοθετεί σε ταχύτατο χρόνο και μέσα σε τρεις ημέρες ψηφίζει νομοσχέδια 500 σελίδες και λύνει όλα τα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και να πω και στην Επιτροπή ότι όταν η Επιτροπή ω Τρόικα ενεργεί και πιέζει την κυβέρνηση εφαρμόζονται. Εδώ τώρα που έχουμε μια νομοθεσία που αν εφαρμοστεί θα είναι υπέρ των πολιτών βλέπουμε και μια δράνεια από την Κομισιόν επί ένα έτος και πλέον διότι από το 2017 έχει έρθει απάντηση και απλά συζητάμε την ελληνική κυβέρνηση ποια θα είναι η αρμόδια επιτροπή να ελέγξει. Θεωρώ λοιπόν ότι απλά κοροϊδεύονται στην, ε, σε αυτό το επίπεδο και η Κομισιόν και η ελληνική κυβέρνηση πετάει ο ένα τον παλάκι στον άλλον και περνάει ο καιρό. Άρα λοιπόν πρέπει να κληθεί η ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η αρμόδια αρχή για να ελέγξει όλο το θέμα. Όμω, επί τη ουσία έχουμε τα εξή ζητήματα. Επιβάλλονται υπέρογγε ε, χρεώσεις εκ μέρους των τραπεζών. Παραδείγματος χάρη το POS. Το POS έρχεται η ελληνική κυβέρνηση με εντολή της Τρόικας και λέει θα το εφαρμόσουν και θα το βάλουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και αν δεν το βάλουν έχουν χίλια ευρώ πρόστιμο και αν δεν το εφαρμόσουν άλλο πόσο πρόστιμο. Όταν λοιπόν λειτουργήσει το POS, το ερώτημα είναι πόσο της εκατό χρέωση θα πάρει η τράπεζα. Διότι αν εσείς είστε ένας δικηγόρος και χρεώσετε κάποιον 500 ευρώ, και πληρώσετε προμήθεια 3-4-5% έχει μεγάλη σημασία. Οι χρεώσεις λοιπόν που επιβάλλουν στη λειτουργία του POS οι τράπεζες είναι υψηλότατες. Και πλέον στα μικρά μαγαζιά, στα περίπτερα, δεν τους συμφέρει να έχουν POS, διότι το κέρδος που βγάζουν πουλώντας τσιγάρα είναι λιγότερο από το ποσοστό που θα πληρώσουν στις τράπεζες. Διότι το κέρδος που έχεις πουλώντας σιγάρα είναι 2% ας πούμε και το ποσό που θα πληρώσεις στην τράπεζα με, λόγω του POS μπορεί να είναι 4%. Επομένως έχεις και ζημία. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεύτερον, επέβαλε η κυβέρνηση να πληρώνεται ο φόρος, η δυσβάστακτη φόρη στην Ελλάδα μέσω τραπεζών και όταν πηγαίνεις στον Κισέ σου ζητάει 2 ευρώ για να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος. Έχουμε τέτοιες χρεώσεις απίθανες. Έχουμε άλλες υπερβολικές χρεώσεις σε σχέση με τις πιστοτικές κάρτες που αναφέρθηκε η Κομισιόν. Έχουμε την απίθανη χρέωση της εισφοράς 128 του 75 που είναι ποσά τα οποία επιβάλλονται ως ε, εισφορές επί των επιτοκίων και υποτίθεται ότι αυτά θα πήγαιναν τα χρήματα για την ενίσχυση των εξαγωγών. Όμω απαγορεύεται η ενίσχυση των εξαγωγών. Και όμω επί 40 χρόνια εισπράττονται αυτά τα ποσά, τα οποία πηγαίνουν πού. Άρα λοιπόν έχουμε, για να κλείσουμε κυρία Πρόεδρε, εδώ τις τράπεζες να είναι κράτος σε κράτη, να επιβάλλουν όποιο ε, ό,τι χρεώσεις θέλουν και να έχουμε μια καταχρηστική λειτουργία. Έχουμε δύο επίπεδα. Έχουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και έχουμε και την καταχρηστική λειτουργία των τραπεζών που επειδή εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες περίπου την ίδια πρακτική στην ουσία έχουν δημιουργήσει concerted practice η οποία εναρμονισμένη πρακτική δηλαδή η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 85 και άρθρο 86 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν διασωθεί με χρήματα του ελληνικού λαού από τα μνημόνια και στο τέλος υφίστανται όλες αυτές τις επιβαρύνσεις και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Πρέπει να πληρώνονται τώρα οι μισθωτοί μέσω τραπέζης. Ξέρετε ότι όταν αποστείλει ο εργοδότης το μισθό στην ε, ε, στο λογαριασμό του μισθωτού πληρώνει ο μισθωτός, τελειώνω, 2 ευρώ. Και δεν μπορεί να ανοίξει ο μισθωτός και νέο λογαριασμό. Άρα λοιπόν εδώ πρόταση. Τι πρέπει να γίνει. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταλεί μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες για καταχρηστική λειτουργία. Δεύτερον, να σταλεί επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η αρμόδια αρχή που ελέγχει τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα. Τρίτον, να σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο έχει αρμοδιότητα για την προστασία των καταναλωτών. Πέμπτον, να σταλεί επιστολή στην ΜΕΑ, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, για το τι επιτέλους θα γίνει και ποια θα είναι η αρμόδια αρχή και να μας πει και η Κομισιόν σε πόσο χρονικό διάστημα προτίθεται να παραπέμψει την Ελλάδα για παραβίαση της νομοθεσίας εάν δεν προσδιορίσει την αρμόδια αρχή που θα ελέγχει την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή και θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση είναι ανοιχτή όπως και άλλες υποθέσεις που σύντομα θα σας έρθουν κυρία Πρόεδρε για την καταχρηστική λειτουργία των τραπεζών και θυμόσαστε είχαμε υποβάλει μια πρόταση να είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη, δεν έγινε δεκτό αυτό, όχι με ευθύνη δικιά σας. Άλλη καταγγελία του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος πάλι για τον τρόπο λειτουργία των τραπεζών σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό θέμα αυτό και απαράδεικτο. Απαράδεικτο αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ε, κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο, ο αναφέρον, όπως πολύ σωστά και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και ο συνάδελφος είπε, κάνει λόγο στην αναφορά του για τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα από τις 28 Έκτου του 2015 και που οδήγησε αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών να συναλλάσσονται με κάρτες και μέσω ποιεώς και ότι με αυτή την αφορμή οι εμπορικές τράπεζες χρεώνουν υπέρμετρες προμήθειες τις οποίες οι επιχειρήσεις λιανικές δεν μπορούν να σηκώσουν, οι οποίες πολλές φορές ξεπερνούν και το 3%. Δεν θα με ακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι καλύφθηκα από τον, τον συνάδελφο, ε, υπόθηκαν τα περισσότερα. Αυτό που θέλω να πω και που πρέπει να προσέξουμε είναι εκτό των άλλων ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, διότι λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει την διαφάνεια και την, ε, και θα ελέγξει και την φοροδιαφυγή. Ε, ε, όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό που γίνεται και που είναι φανερό πια είναι το γεγονός ότι με αυτή τη διαδικασία ακριβώς μεγιστοποιεί τα κέρδη των ε, ελληνικών τραπεζών. Ε, και ενώ πιέζει τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο ε, συναλλαγής, την ίδια στιγμή το ίδιο το κράτος δεν προστατεύει τους πολίτες από τα αποτελέσματα αυτής της συναλλαγής. Με υποχρεώνει δηλαδή να, μέσω των capital control να κάνω τέτοιου είδους συναλλαγή, όμως η αρμοδιότητα που ανήκει αυτή τη στιγμή στο κράτος, που είναι ο έλεγχος των τραπεζών, δεν το κάνει, που είναι ο έλεγχος της φοροδιαφυγής, το ελληνικό κράτος δεν το κάνει, το χρεώνει στον πολίτη δηλαδή η τράπεζα μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Ε, νομίζω ότι, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, όχι να, ε, νομίζω, είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αυτή αναφορά, ε, και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόρο για τον ίδιο τον πολίτη, δεν μπορεί να κάνει συνεχώ αναφορά, ούτε μπορεί να έρχεται εδώ πέρα. Προτείνω να ζητήσουμε μια λεπτομερή αναφορά για το καθεστώ των τραπεζών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στι προσωπικέ προσπάθειε που έκανα για να μπορέσω να μάθω τι ακριβώ γίνεται, ποιε είναι οι συναλλαγέ, δεν μπόρεσα να μάθω απολύτω τίποτα. Θα περίμενα φυσικά να υπάρχει μια, μια λίστα τιμών. Να ξέρουν οι πολίτε ποιο, ποιο ακριβώ είναι το κόστο τη ε, της συναλλαγής τους. Και αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ε, ό,τι υπάρχει είναι αποτέλεσμα των προσωπικών συναλλαγών που γίνονται μεταξύ του πολίτη και της ε, τράπεζα. Και επειδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να εξαδίωσουμε το θέμα στο ότι πήραμε μια απάντηση από την Επιτροπή και τελειώσαμε με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί πιστεύω πραγματικά και εγώ ότι αγγίζεται τα, τα όρια της εσχροκέρδειας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε ίσως και κάποια πρωτοβουλία. Να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να προτείνει ε, κάποιες θέσεις οι οποίες να τίνουν προς την κατέθεση του ελέγχου αυτής της κατάστασης. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, για, την συνεισφορά σας και για την, μάθημα. Λοιπόν, δεν έχω... I don't have any, any, any Δεν έχω κάποιον άλλο στο κατάλογο των ομιλητών σήμερα. Ό αναφέρον απουσιάζει. Είμαι βέβαιη ότι μαζί με την Κομισιόν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για αυτή την αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα μείνουμε σε στενή επαφή. Θα ήθελα να σας παροτρινώ να επιδιώξετε λίγο περισσότερο να βρούμε μια εξήγηση, μια λύση όσον αφορά το μην καθορισμό της αρμόδιας αρχής και όσον αφορά και την ελληπή επικοινωνία των ελληνικών αρχών. Σας παροτρύνω λοιπόν να το δείτε αυτό το θέμα και να επανέλθετε να μας απαντήσετε με κάποια επιστολή αν έχετε μια απάντηση και εμείς ε, θα πρέπει να στείλουμε μια επιστολή εκ μέρους της Επιτροπής της Αρμόδιας Αρχές δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομίας, στην ε, Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού κτλ. Ρωτώντας για ποιο λόγο χρειάζεται τόσο χρόνος για να διοριστεί κάποια αρχή και να δούμε και πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν ε, την όλη έρευνα, πώς θέλουν δηλαδή να προχωρήσουμε όσον αφορά αυτή την ε, καταγγελία. Επ' αυτού πιστεύω μπορούμε να συμφωνήσουμε κύριε Μαριά. Να μπούμε στο ελεγκτικό μέρος. Δηλαδή, εδώ έχουμε καταγγελία για καταχρηστική λειτουργία των τραπεζών. Στην Ελλάδα έχουμε δύο ειδών τράπεζες αυτές που ονομάζονται συστημικές τράπεζες, δηλαδή είναι τέσσερις μεγάλες τράπεζες και αρμόδιο όργανο, αρμόδια, αρμόδια αρχή για να τους ελέγξει είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το σύστημα ε, και η κυρία Νουή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει εκεί η επιστολή. Για τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες, γιατί είναι αρκετές άλλες, αρμόδια, αρμόδια αρχή που ελέγχει όλα αυτά είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Επομένως οι επιστολές πρέπει να γίνουν και στις εποπτικές αρχές των τραπεζών. Η μία περίπτωση είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες και η άλλη είναι η Τράπεζα της Ελλάδος για τις υπόλοιπες μικρές εμπορικές τράπεζες. Διότι εδώ έχουμε καταχρηστική λειτουργία των τραπεζών. Ε, Νομίζω ότι θέλω να παραμείνουμε σε αυτά που πρότεινα. Δεν είναι δική μας υπόθεση να κάνουμε διάκριση μεταξύ διαφόρων τραπεζών. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης να το κοιτάξει. Να θέλω να διαφωνήσω. Ένα πράγμα είναι η ελληνική κυβέρνηση με τον οργανισμό που θα φτιάξει να έχει την ευθύνη εφαρμογής του κανονισμού και ένα άλλο πράγμα είναι η καταχρηστική λειτουργία των τραπεζών που αυτό ελέγχεται από τις εποπτικές αρχές των τραπεζών και εν προκειμένου στην Ελλάδα είναι δύο οι εποπτικές αρχές τραπεζών. Η ECB, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλάδος για τις υπόλοιπες. Να στείλουμε και εκεί επιστολές για να αναγκαστούν να συμμορφωθούν. Ωραία, ας προχωρήσουμε έτσι να δούμε αν θα μας απαντήσουν. Αλλά και τους υπόλοιπους που σας είπα, οπωσδήποτε θα πάρουμε απάντηση. Ωραία. Άλλη μια επιστολή να στη στείλουμε. Εμείς είμαστε μέγας επιστολικός ε, φίλος στην Ευρώπη, γιατί έχουμε αλληλογραφία με πολύ κόσμο. Λοιπόν, 8. Διευθυντική επίσκεψη στη Λάρνακα, Κύπρος. Επικεφαλής αντιπροσωπείας περιέργως ο κύριος Τσάκη, ο οποίος αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη για τη λειτουργία και την επικοινωνία αυτής της Επιτροπής και τη φέρνει σε πέρας αξιοθαύμαστα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα η κατάσταση έχει ως εξή. Ήταν πολύ καλή η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή και η επίσκεψή μας στην Κύπρο. Ήταν εξαιρετική προετοιμασία οφείλω να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η συνεργασία ε, με τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν αγαστή επίσης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Η έκθεση εκπονείται αυτόν τον καιρό. Πολύ σοβαρή και πολύ καλή και σας ευχαριστώ για τη σύνταξή της. Κοιτάξτε τώρα, το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σοβαρό. Υπάρχει ένταση ανάμεσα στο Δήμο της Λάρνακας και το λιμένα της Λάρνακας, διότι έχουν διαφορετικά συμφέροντα και επίσης υπήρχε και έλλειψη διαλόγου. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Όπως και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές δεν συζητούσαν με τη συγκεντρική κυβέρνηση, τα υπουργεία. Αρχίσαμε λοιπόν ένα καλό διάλογο. Ε, μεσολαβήσαμε δηλαδή να αρχίσουν να συζητάνε ο Δήμαρχος με το Λιμένα ε, το πρόβλημα ε, ποιο είναι. Το λιμάνι είναι σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία δίπλα στη Λάρνακα και φυσικά καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργούνται εντάσεις και προβλήματα. Άλλα συμφέροντα έχει η πόλη και η περιφέρεια λόγω τουρισμού και άλλα συμφέροντα έχει το λιμάνι. Έχει κάποιες λιμενικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με όλα αυτά και μερικές εταιρείε που δραστηριοποιούνται εκεί έχουν άλλα συμφέροντα του λιμανιού. Το πιο σημαντικό που είχαμε και ως συζήτηση ήταν ε, μια συνομιλία με το Υπουργείο Οικονομικών που μας είπε ότι τελείωσαν την προετοιμασία και το σχεδιασμό για να φτιαχτεί ένα λιμάνι έξω από την πόλη. Αυτό είναι καλή λύση και για τον ίδιο το Δήμο της Λάρακας και για τις εταιρείες αυτές τις ε, εμπορικές ε, στο λιμένα της Λάρακας. Ελπίζω λοιπόν να είναι χρήσιμο το έγγραφό μας και η πολιτική δραστηριότητα για τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Λάνακας. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τη δράση τους και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Υποστηρίζουμε τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα στεναρά από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ήθελα να σας συνειδητοποιήσω συνάδελφοι πως ε, κάποια μέλη... Α, ωραία. Ήρθε και η Άγχελα. Νομίζω μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια και θα ήθελα να σε καλωσορίσω κιόλας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως πρέπει να δώσουμε ένα θετικό πρόσημο σε αυτή την έκθεση που παρουσιάσουμε σήμερα γιατί η γραμματεία ε, μόλις γύρισε από την Κύπρο έκανε επαφές με τα μέλη της αντιπροσωπείας για να λάβει υπόψη τι είχαμε να πούμε εμείς και τα έβαλε στην έκθεση. Τους ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ επίσης και το υπόλοιπο ε, των μελών της αντιπροσωπείας γιατί όλοι έλαβαν υπόψη τα όσα είπαμε εμείς για τα συμπεράσματα. Θα ήθελα επίσης να αξιολογήσω θετικά την δέσμευση που εξέφρασαν οι Κυπριακές Αρχές έτσι ώστε το λιμάνι της Λάρνακας να, περιορίσει, να περιοριστεί σε εμπορικές και τουριστικές ε, δραστηριότητες και να μην συνεχίσει η εκβιομηχάνηση και οι πετρελαϊκές ε, δραστηριότητες να μεταφερθούν εκτός Λάρνακας. Παρόλα αυτά στην έκθεση είναι πολύ σαφές πως αυτή είναι η θέληση μεν των, Κυπριακών αρχών αλλά στο λιμάνι της Λάνακας πρόσφατα ανανέωσαν τις άδειες λειτουργίες πετρελαϊκές εταιρείες και δεν έχει ε, ημερομηνία λήξης αυτή η ανανέωση. Οπότε αυτό έρχεται σε κάποια αντίφαση με τις δεσμεύσεις για μεταφορά των εγκαταστάσεων που έχουν ακουστεί. Οπότε θα πρέπει εμείς στην Επιτροπή Αναφορών να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθήσουμε το θέμα. Θέλω να τονίσω επίσης πως οι διατάξεις της Σύμβασης Σαρούς έχουν καταπατηθεί και οι εκ των υστέρων συναντήσεις ενημέρωσης ε, των Κυπριακών Αρχών δεν βοήθησαν στο να συμμορφωθούμε με τη σύμβαση, δεν συμβάστηκαν την υποχρέωση να ενημερώνουν το ε, κοινό, όπως επίσης και οι προθεσμίες δεν έγιναν σεβαντιστές. Μία προσπάθεια μυστικοπάθειας θα έλεγα, ε, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα όσα ήθελαν να κάνουν τοπικές αρχές και το Δημαρχείο. Και όπως μας είπαν οι αναφέροντες, τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ νέου που μας κοινοποίησαν όλα αυτά τα στοιχεία, ο κίνδυνος για ατυχήματα εξακολουθεί να υπάρχει. Παρόλο που είναι μόνο ε, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου ε, παρόλα αυτά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό και ο κίνδυνος υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ, οι συστάσεις σας είναι σωστές και θα πρέπει να σας ενημερώσω πως εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες αλλά όχι κάτι το σημαντικό. Και ήταν μια πολύ ικανοποιητική αποστολή πρέπει να πω. Ωραία, χαίρομαι που ήταν επικοδομητικό το ταξίδι αυτό και που συμφωνούμε όλοι. Επ' αυτού ο κύριος ε, Σόλτ επίσης ήταν και μέλος της αντιπροσωπείας, θέλετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου και ειδικότερα τη γραμματεία για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου έκθεσης αποστολής ε, και τη σύσταση. Ήθελα να πω ότι πέραν ε, των ε, σχολείων που μόλις ακούσαμε θα ήθελα να προσθέσουμε κάποιο κείμενο στα τελικά συμπεράσματα. το οποίο θα αφορά κάποια σημαντικά θέματα. Την έλλειψη της ε, περιβαλλοντικής ε, εκτίμησης ε, που είναι σημαντική σε τέτοιες περιπτώσεις. Και θα χρειαστεί να προσθέσουμε και άλλο κείμενο το οποίο θα αφορά την ε, πραγματική φύση της ε, δράσης ε, από τον αναφέροντα και το τελευταίο θα κάνει μια γενική αναφορά στις κύριες πτυχές που θα αφορά ένα από τα βασικά θέματα της αναφοράς θα στείλουμε τα σχετικά κείμενα στη γραμματεία με τις παρατηρήσεις μας. Θα τους πούμε και πού πρέπει να μπει αυτό το κείμενο, πώς θα ενσωματωθεί στο τελικά συμπεράσματα και τις συστάσεις. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τη γραμματεία. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς κύριε Σόλτες. Και η Κομισιόν εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Παρζάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια. Διάβασα την έκθεση και θεωρώ ότι η αποστολή αυτή υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και οι συστάσεις είναι εξαιρετικές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλες αυτές τις προσπάθειες. Πρόεδρο, ευχαριστούμε και για τη δική σας συμβολή μέχρι στιγμής. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, όπως βλέπω. Να σας υπενθυμίσω τώρα ότι η προθεσμία για τροπολογίες τροπολογίες ε, που μπορείτε να κάνετε μόνο για το κομμάτι των συστάσεων η, δεύτερη 2η Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι είναι η προθεσμία μετά από εκείνη τη χρονική στιγμή θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 21 Φεβρουαρίου σε μια συνεδρία της Επιτροπής. Αυτά. Και εδώ κλείνουμε για σήμερα. Το οποίο σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία να πάτε πίσω στα γραφεία σας, να κάνετε κάποια γρήγορα τηλεφωνήματα που επήγουν και να ξανάρθετε για το κοκτέιλ στο εστιατόριο των μελών, στο σαλόνι Αριθμό 4. Όλοι είναι καλεσμένοι, ειδικότερα η Κομισιόν, από τις 6 και 4. Κάντε γρήγορα τα τηλεφωνήματα που έχετε να κάνετε και φύγαμε και θα συνεχίσουμε για όσο θα υπάρχει κόσμος και ποτά και σνακ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε λιγάκι.